Βαλέντσα παρουσίασε το σχέδιο γνωμοδότησής του, σύστασής του, κατετέθησε μονάχα μία τροπολογία μέχρι το Σεπτέμβριο που ήταν η προθεσμία τροπολογιών από τον ίδιο τον εισηγητή. Εκτός αν ο εισηγητής λοιπόν θέλει να πει κάτι μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Έχετε τις κάρτες σας ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Προχωρούμε λοιπόν κατευθείαν προς την ψηφοφορία. Τροπολογία 1 για την παράγραφο 1 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Γιατί όχι. Ο κύριος Σαλάτο έβαλε ανάποδα την κάρτα του. Τώρα εντάξει. Ψηφίσατε όλοι οι άλλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ομόφωνα εγκρίνεται αυτή η τροπολογία. Συγχαίρω τον εισηγητή. Και τώρα η ψηφοφορία του σχεδίου ψηφίσματος, νομοθετικού ψηφίσματος ως σύνολο, άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, ψηφίσατε όλοι. Όχι ακόμα, δεν ψηφίσατε όλοι. Α, εγώ ξέχασα να ψηφίσω, όλοι από όλους. Πέρασε. Πάλι ομόφωνα εγκρίνεται και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο Βαλέντσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στο σημείο 6, εταιρική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσων του Σολομώντα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Πετραουνέβης. Πρόταση ε, που βασίζεται επίσης στο άρθρο 201.6. Ζητείται η σύμφωνη γνώμη μας και η έκθεση αυτή δόθηκε στην κυρία Πετραουνέβης από την ομάδα του ΕΛΚ Στι 2 Ιουλίου η Κομισιόν παρουσίασε την πρότασή τη και η συγγήτρια παρουσίασε το σχέδιο του γνωμοδότησής τη στι 14 Ιουλίου. 2 Σεπτεμβρίου ήταν η προθεσμία για τι τροπολογίε. Πέντε τροπολογίε κατατέθηκαν, μία εκ των οποίων θεωρήθηκε μονάχα παραδεκτή από την Πρόεδρό μας μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες επιτροπές. Πήραμε τροπολογίες επίσης από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Όπως ξέρετε, βάσει του κανονισμού του Κοινοβουλίου, στην ειδική αυτή διαδικασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του ή να αρνηθεί τη σύμφωνη γνώμη του σε σχέση με την Διεθνή Συμφωνία την εν λόγω και μόνο περιορισμένες αιτήσει διαδικαστικού χαρακτήρα μπορούν να προσθεθούν στο νομοθετικό ψήφισμα μετά από ένα ενδελεχή έλεγχο της ε, του αποδεκτού, του παραδεκτού αυτών των ε, εκθέσεων. Και έχει γίνει αυτός ο έλεγχος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκτός αν θέλει να πει λοιπόν κάτι η συγγήτρια, όχι λέει αρνητικά η συγγήτρια, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για την έκθεση της κυρία Πετράου Νέβης. Τροπολογία υπαριθμών 3, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Ομόφωνα δεκτή. Ψηφοφορία στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ως σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορία. Και πάλι ομόφωνα και συγχαίρω την κυρία Πετραουνέβη. Το σημείο 7 τώρα, όπως είπα προηγουμένως, αναβλήθηκε και θα εξεταστεί προηγουμένως από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σημείο 8, έλεγχος και αστυνόμευση για την περιοχή που καλύπτεται από τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον Βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό. Πρόκειται για μια πρόταση τροποποίησης και ενημέρωσης των κυρωτικών κανόνων που περιλαμβάνει το σύστημα εποπτείας το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή Αλίας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Καμία πολιτική ομάδα δεν έχει ζητήσει να πάρει αυτή την έκθεση και ως αποτέλεσμα η κυρία Κάρμεν Φράγκα ως πρόεδρος της ε, Επιτροπής Αλίας ανέλαβε την έκθεση αυτή. Το αρχικό σχέδιο παρουσιάστηκε στις 3 Νοεμβρίου. 5 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους ήταν η προθεσμία για τροπολογίες. Τρεις τροπολογίες είχαν κατατεθεί μέχρι τότε η πρόταση αυτή παρεπέμφθη από, το, από την προηγούμενη ε, Επιτροπή βάσει της διαδικασίας διαβούλευσης πριν από τη θέση εφαρμογή της Συνθήκης Λισαβόνας, αλλά μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας που σε εφαρμογή, είχαμε αποφασίσει να ζητήσουμε πολιτική εντολή για να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου και τώρα υπόκειται στην συναπόφαση. Οι διαπραγματεύσεις αφορούσαν τα θέματα των πολλαπλών ενημερώσεων πολλών άρθρων που έχουν να κάνουν με την επιτροπολογία για να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης, η προσαρμογή του τελικού κειμένου που είχε εγκριθεί θα πρέπει να γίνει. Επετεύχθη τελικά <clears throat> στον τριγωνικό διάλογο που είναι στις 15 Σεπτεμβρίου για να υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο πρώτη ανάγνωση και αυτό το κοινό κείμενο συμφωνίας θα πρέπει να υποβληθεί σε επίσημη ε, ψηφοφορία από την Επιτροπή μας ως μια επίσημη νομοθετική τροπολογία και μετά από διαβούλευση με την ΚΟΡΕΠΕΡ θα έρθει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αποτελέσει την οριστική συμφωνία. Το κείμενο της οριστικής συμφωνίας, εάν δεν υπάρχουν λοιπόν καθόλου αντιρρήσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με τη συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα. Και αυτό σημαίνει ότι όλες οι άλλες ε, τροπολογίες καταπίπτουν. Και πάμε στην ε, νομοθετική πρόταση ως τροποποιηθήκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίνεται ομόφωνα και κατόπιν έχουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε. Εγκρίνεται ομόφωνα, τα πάμε πάρα πολύ καλά σήμερα το πρωί. Ε, συγχαίρω λοιπόν την κυρία Φράγκα, την πρόεδρό μας. Ομοφωνία λοιπόν. Σημείο υπαριθμών η Τροποποίηση του κανονισμού 2187 κάτω 2005 του Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση διαλογής αλληλευμάτων ανώτερη κατηγορίας και του περιορισμού αλλιές όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι στα έντατα τη Βαλτική θάλασσα, των Μπέλτ και του Σάουντ. Εδώ ε, προτείνεται να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Συμβουλίου που ορίζει συγκεκριμένα ε, μέτρα για την αλία στην ε, Βαλτική, των τον και του Σάουντ. Αναφέρεται το, τα είδη, το μέγεθος και οι περιοχές των ψαριών και οι τροπολογίες που θα συμπεριληφθούν από το 2011. Εκεί προβλέπονται κάποιες ε, διατάξεις που ε, αφορούν στην, στον περιορισμό της αλίας, κανονισμός ε, του 2009 που ορίζει τις δυνατότητες αλίας για συγκεκριμένα είδη ψαριών που υπάρχουν στη Βαλτική θάλασσα και κανονισμοί που ισχύουν στη Βαλτική για το 2010. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας είναι απαραίτητο τα τεχνικά μέτρα να βγαίνουν από το νομοθετικό πλαίσιο και επιπλέον επειδή ε, είναι τα μέτρα αυτά ε, μόνιμης εφήσεως. Ε, η έκθεση είναι του κυρίου Γκρομπάτσεκ. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου η Επιτροπή παρουσίασε τις απόψεις της. Σήμερα ο κύριος Γκρομπάτσεκ θα παρουσιάσει το δικό του το σχέδιο έκθεσης και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκρομπάτσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή, δεν κατατέθηκαν τροπολογίες. Δύο σχόλια μόνο έχω να κάνω και δυστυχώς ε, τα έχω ξαναπεί και πρέπει να τα επαναλάβω. Το ένα αφορά την ε, ποιοτική επιλογή για τα ίδια αυτά στη Βαλτική θάλασσα. Είναι λογική η πολιτική για απαγόρευση των απορρίψεων. Θα ήθελα ωστόσο να σας μιλήσω για την κατάσταση σε σχέση με τα δύο αυτά η τη χωματίδα και το καλκάνι δηλαδή, αλλά και για τον γάδο. Στην περίπτωση της χωματίδας, που αλλιεύεται την άνοιξη, τους αριουνούς μήνες, η αλληλεία στη Βαλτική γίνεται λίγο πολύ με βάση τους ισχυόντες κανόνες. Η χωματίδα που αλλιεύεται κατά τις αριθμούς μήνες, όπως είπα, δεν έχει καμία εμπορική αξία. Επομένως, είναι χάσιμο χρημάτων το να την αφήνεις ε, στο κατάστρωμα του σκάφους, να τη μαζεύεις. Και εξού η απόρριψή της στη θάλασσα. Η χωματίδα εφόσον ξαναρριχθεί στη θάλασσα ζει, δεν πεθαίνει όπως ο γάδος. Άρα, απαγόρευση των απορρίψεων χωματίδας και καλκανιού με βάση αυτό που σας προείπα είναι κάτι που δεν έχει λογική. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ την Επιτροπή, από την Επιτροπή να το ξαναεξετάσει. Βέβαια, η έκθεση δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία για την απαγόρευση των απορρίψεων. Αν όμως ακολουθήσουμε μια γενική προσέγγιση, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ χειρότερα. αν είναι γενική η προσέγγιση για την απαγόρευση των απορρίψεων και όχι ειδική, αναείδος δηλαδή. E, Τώρα τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα οι μικρότερου μεγέθους, μικρότερων διαστάσεων ε, ψαριών δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τα σκάφη τα οποία αλλιεύουν με τη μορφή του fodder fishing. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία και δεν είμαστε βέβαιοι για το κατά πόσον υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ε, παρεμπίμπτοντα αλλιεύματα. Αν προσθέσουμε τον πλήρη, την πλήρη απαγόρευση των απορρίψεων, μαζί με όλα τα άλλα μέτρα, ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι να υποβαθμίσουμε τα αποθέματα, τα αλλιευτικά στη Βαλτική. Το έχω πει, το έχω επαναλάβει και δεν μπορώ να επιμείνω άλλο σε αυτό το θέμα που αφορά τις ε, τα αλλιεύματα που θα χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χωματίδα και σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, το σημείο 26, 28, αυτές οι υποδιαιρέσεις νοτίως του, το να κλείσουν αυτές οι περιοχές, δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικό λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω τα ψάρια δεν προστατεύονται ήδη όπως η χωματίδα παραδείγματι. Η προσέγγιση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιλέγει αυτές τις προστατευμένες περιοχές και αν λάβουμε υπόψη μας την αλλαγή του κλίματος βάσει των στοιχείων που έχουμε από την έρευνα, ε, τουλάχιστον εγώ δεν πείθομαι για τη Βαλτική. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή κύριε Γκρομπάτσουκ. Ο κύριος Βαλένσα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από τη δική μου πλευρά εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν στα πλαίσια της βιολογικής προστασίας των αποθεμάτων. Είναι απαραίτητο να μας εξηγήσει γιατί στις υπερδιαιρέσεις αυτές, αυτές από 26 έως 30 για το καλκάνι, ισχύουν αυτές για το καλκάνι και το, για τη χωματίδα μάλλον και 22 με 24 για το καλκάνι. Αυτά όμως τα είδη, τα θαλάσσια, βρίσκονται σε όλη την περιοχή της Βαλτικής. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα πληρέστερο σχήμα, ένα πληρέστερο σύστημα προστασίας του σε όλη τη Βαλτική. Έχουν τεράστια σημασία για το τοπικό οικοσύστημα της Βαλτικής. Γι' αυτό τα ευρωπαϊκά όργανα που είναι αρμόδια για την αλία θα πρέπει να λάβουν υπόψη σοβαρά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λέβεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ε, ευχαριστώ κύριε Γκρόμπασεκ για τις εξηγήσεις που μου δώσατε. Σε ό,τι αφορά τώρα την απόρριψη των πλατιψάρων, των ε, πλατέων ηχθείων, Δυστυχώς δεν επιβιώνω όλα τα πλατύψαρα τα οποία απορρίπτονται στη θάλασσα. Ακόμα και αν από βιολογική έποψη θεωρητικά μπορούν να επιβιώσουν αντίθετα από ό,τι συμβαίνει πραγματικά με το γάδο με το βακαλάο. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν πολλά θαλασσοπούλια τα οποία παρακολουθούν εντέχνως τα αλλιευτικά πλοία και τα οποία εκμεταλλεύονται αυτές τις απορρίψεις. Γι' αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο στο βαθμό του δυνατού να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο επιλεκτική ε, επιλεκτικά μέτρα σε ό,τι αφορά τις απορρίψεις και να έχουμε τη γενική αυτή η δυνατόν απαγόρευση των απορρίψεων γιατί αλλιώς έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι ανησυχητική στη, Βαλτική. Προ την Κομισιόν, σε ό,τι αφορά τι τεχνικέ αυτέ ρυθμίσει που ισχύουν στη Βαλτική, η δική μου εντύπωση ήταν ότι ορισμένα κράτη-μέλη καταβάλουν προσπάθειες να εισάγουν και άλλε τροποποίησει στις τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν τη Βαλτική, παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά στο Βακαλάο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, <clears throat> ελπίζω ότι το θέμα αυτό θα έλθει και ενώπιον του Κοινοβουλίου και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτές τις ε, προτινόμενες προσαρμογές. Δεν θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να παρακάμπτουν την ε, γνώμη του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Επίσης, σε ό,τι αφορά το καλκάνι, το ερώτημά μου είναι μήπως θα έπρεπε και αυτό να περιλαμβάνεται στα συνολικά αλλιεύματα, όπως προτείνει η Κομισιόν ή όχι. Κύριε Γκρομπάτσεκ, μετά από την Κομισιόν θα σας δώσω το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Κάποια σχόλια θέλω να κάνω, λέει ο κ. Γκρομπάτσεκ. αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως. Δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει από τη δική μου θέση, από τις δικές μου ιδέες. Δεν είναι κάτι που προκύπτει από επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Είναι η άποψη την οποία έχουν εκφράσει οι μικροί αλείς. Πολλές φορές απορρίπτουν την χωματίδα γιατί δεν έχει καμία εμπορική αξία και πιστεύουν ότι μια τέτοια συμπεριφορά ευθυγραμμίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί δεν, έχουν, δεν έχει για αυτούς νόημα το να εκφορτώνουν στα λιμάνια την χωματίδα. Η κυρία Γιοψένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα. Θα ήθελα να, θέσω και, να προσθέσω και το ερώτημα του κυρίου Βαλένσα προς την Κομισιόν. Από ό,τι καταλαβαίνω, όταν τα νέα αυτά τεχνικά μέτρα τα οποία εισήγαγε η Κομισιόν να έρθουν σε εφαρμογή του χρόνου θα περιλαμβάνουν και ορισμένε βασικέ αρχές και το ερώτημα είναι κατά πόσον αποτελεί πρόθεσή σα στην περίπτωση αυτή το σύνολο των τεχνικών αυτών μέτρων να επαφίενται στις περιφερειακές δομές διαχείρισης της ε, αλίας που θα προκύψουν από τη διαδικασία μεταρρύθμισης τη ε, αλληλευτική πολιτική. Δηλαδή, θα υπάρξει περιφερικοποίηση των τεχνικών μέτρων επί τη βάση των γενικών αρχών που έχει θεσπίσει η Κομισιόν ή είναι η πρόθεσή σας να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία επιτροπολογίας για μια πιο λεπτομερή εφαρμογή τεχνικών μέτρων. Γιατί προφανώς είναι διαφορετικές οι δύο προσεγγίσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα μέλη της Επιτροπής μας. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Γεψένα. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή τον εισηγητή για την έκθεσή του και για την αξιολόγηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, φυσικά η όλη νομική δομή και αρχιτεκτονική είναι υποδιαπραγμάτευση στην Επιτροπή αυτή την περίοδο. Ωστόσο, η ιδέα για τα τεχνικά μέτρα βασίζεται στο ότι ναι, υπάρχει ένας γενικός κανονισμός για τα τεχνικά μέτρα. Αλλά έχει ήδη περιφερειοποιηθεί. Όπως βλέπετε, ο κανονισμός για τη Βαλτική αφορά και ισχύει μόνο για τη Βαλτική. Είναι σαφές ότι διαφορετικά ύδατα, διαφορετικά αλλιεύματα. Χρειάζονται διαφορετικά μέτρα. Δεν μπορούν να καλυφθούν όλα από έναν και μόνο κανονισμό. Όπως έδειξε επίσης η εμπειρία μας, χρειάζεται μια διαδικασία για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να τροποποιούμε τις διαδικασίες αυτές, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιες περιβαλλοντικές αλλαγές και αλλαγές ε, στις επιστημονικές συμβουλές. Τώρα, πώς ακριβώς ε, θα είναι η τελική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι θα περιέχει, δεν μπορώ να το προδικάσω από τώρα. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κ. Βαλένσα, θα πρέπει να επανέλθω να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Πώς δηλαδή εμφανίστηκαν ε, αυτές οι διατάξεις, ιδίως για τον κανονισμό των ετήσιων ε, τάξ, ό,τι αφορά την ε, συγκεκριμένη ε, περιοχή, τη Βαλτική θάλασσα. Νομίζω ότι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Βαλτικής θάλασσας, που δημιουργήθηκε μετά την τελευταία διεύρυνση του 2004. Αυτές οι διατάξεις μεταφέρθηκαν από την απόφαση της αποφάσεις της Επιτροπής αυτής στον κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα που αφορούσαν τη Βαλτική. Θεωρήθηκε ότι ήταν ε, ο πιο εύκολος τρόπος. Βέβαια δεν έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής με τα κράτη-μέλη το εύρος στο πεδίο εφαρμογή της ρήτρα αυτής για το καλκάνι και για τη χωματίδα. Θα μελετήσουμε λοιπόν το ερώτημά σας. Θα ζητήσουμε από τους επιστήμονες να εκτιμήσουν ε, αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής ε, των περιοχών αυτών στο μέλλον. Γιατί όχι. Αυτά είχα να σας πω. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος και εμείς σας ευχαριστούμε. Μήπως ε, ε, θέλετε εσείς ε, να λάβετε και πάλι το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ένας εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν είπε ότι το θέμα αυτό ε, συζητήθηκε κατά την πρώτη μας συνάντηση, τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε η έκθεση. Και τότε λοιπόν μας είπαν ότι υπάρχουν οι μελέτες και με βάση αυτές τις μελέτες ορίστηκαν οι κλειστές περιοχές. Τελικά τι γίνεται, υπάρχουν οι μελέτες ή όχι. Και ποιος αποφασίζει Ποιε περιοχές είναι κλειστέ και προστατεύονται και ποιε όχι. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στις κλειστέ περιοχές τα αλλιεύματα χωματίδας ανέρχονται σε περίπου 100.000 τόνους. Όσον αφορά τις απροστάτευτες περιοχές, εκεί μιλάμε για χίλιους τόνους. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει περιθώριο συζήτησης και νομίζω ότι χρειαζόμαστε πληροφορίες για τη βάση πάνω στην οποία παίρνει η Κομισιόν τις αποφάσεις της. Παρακαλώ, κυρία Λόβα. Η εντύπωση. Να πω το εξής. Ε, η Κομισιόν δεν μου απάντησε. Εγώ ρώτησα κατά πόσον ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να συζητήσουν και για άλλα είδη ψαριών ε, σε σχέση με αυτόν τον κονισμό. Παραδείγματο χάρη σε σχέση με τον βακαλάο. Ε, κατώτατα τάκ. Θα συζητηθεί αυτό. Ε, ζητώ συγγνώμη, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τι ακριβώς ε, εννοείται με τη συζήτηση άλλων ειδών ψαριών. Για απαγόρευση μιλάτε. Μήπως μπορείτε να εξηγήσετε. Τι ακριβώς ρωτάτε. Κοιτάξτε, εγώ πήρα την εξή πληροφορία, ότι στον Βακαλάο θα μειωθεί το κατώτατο όριο. Και στόχος είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν ε, μικρότερες απορρίψεις. Θα μειωθεί το λιγότερο ελάχιστο βάρος αλλά δεν είναι ότι αυτό αναφέρεται στον κανονισμό. Γι' αυτό λοιπόν ρώτησα την Κομισιόν και τα κρατημέλη κατά πόσον θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Βεβαίω ε, ζητώ συγγνώμη. Δεν, είχα, δεν έχω μπροστά μου τα πλήρη πρακτικά για το τι ελέγχθη ε, στην προηγούμενη συζήτηση. Όσον αφορά το βακαλάο, Ε, συζητήθηκε αυτό στην ε, ομάδα εργασίας όσον αφορά το φύλλο που πρέπει να ακολουθήσουμε σχετικά με τις απορρίψεις όπως πρότεινε και το Συμβούλιο ε, πέρυσι το Συμβούλιο του Οκτωβρίου κάλεσε την Κομισιόν να καταρτήσει ένα είδος χάρτη αποφυγής απορρίψεων. Και υπήρξαν κράτη-μέλη που πρίτειναν το ελάχιστο μάγεθος εκφόρτωσης. Ε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό συζητήθηκε σε βάθος ε, ε, εκ μέρους των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν προτείνουμε αλλαγές στο ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης. Είναι σαφές αυτό και με ανακουφίζει αυτό που λέτε, διότι όπως ξέρετε οι βακαλάοι αρχίζουν να αναπαγωγεί στα 4-5 χρόνια μονάχα. Άμα μειώσει κανείς το ελάχιστο βάρος το μέγεθος της εκφόρτωσης. Αρχίζει κανείς και εκφορτώνει ε, νεαρούς βακαλάους, οι οποίοι δεν είναι ακόμα σε ηλικία αναπαραγωγής. Αυτό σε εποχή που υπάρχει μεγάλη πίεση στα αλλιευτικά αποθέματα. Δεν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Αν δεν θέλει να επανέλθει ο κύριος Γκραμπάτσεκ, πρέπει να σας πω ότι η προθεσμία των τροπολογιών για αυτή την έκθεση είναι η 5η Οκτωβρίου, 12 <clears throat> μεσημέρι και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 26 και 27 Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο. Εφόσον συμφωνούμε λοιπόν με αυτές τις ημερομηνίε μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης ενδιάμεση εταιρικού χαρακτήρα συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και χωρών του Ειρηνικού. Η συγγήτρια για την έκθεση αυτή ήταν η κυρία Φράγκα. Τώρα, ζητάτε η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για να μπορέσει να συναυθεί πλήρως η συμφωνία αυτή βάσει του άρθρου 201.6. Η... Το θέμα αυτό έχει παραπευθεί στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που έχει τον κύριο Ντέβιτ Μάρτεν ως εισηγητή. Η δική μας Επιτροπή αποφάσισε να γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό και η κυρία Φράγκα η πρόεδρο μας έχει αναλάβει τη γνωμοδότηση αυτή. Η Κάρμεν όμως δεν είναι παρούσα σήμερα. Ζήτησε από τον Αλέν Κάντεκ να παρουσιάσει αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση εκ μέρους της. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Καντέκ και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση με τα άλλα μέλη και μπορούμε να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν σχετικά. Ο Αλάν. <coughs> Σας ευχαριστώ. Πρόκειται απλώ για μια γνωμοδότηση, μεν, αλλά πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό αυτό ο φάκελο για ορισμένα ολιστήματα της Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει προετοιμάσει μια έκθεση για τη σύναψη μιας εταιρική οικονομική σχέσης, η οποία ισχύει προσωρινά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της, του Ειρηνικού Νέα Γουινέα, νήσι Φίτζη. Πρόκειται για μια έκθεση που υπόκειται σε διαδικασία σύμφωνη γνώμη με συγκριτή τον κύριο Ντέβιτ Μάρτιν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόεδρο μα, η κυρία Φράγκα, ήθελε η Επιτροπή Αλία να δώσει μια γνωμοδότηση η οποία να προσανατολίζεται προ του κανόνε προέλευση για τα προϊόντα αυτά σε ό,τι αφορά τον τόνο που αλλιεύεται στι χώρε αυτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πράγματι δασμολογικέ προτιμήσει για ορισμένα προϊόντα και ιδίω στι κονσέρβες τόνου, με την προϋπόθεση ότι είναι πράγματι προερχόμενα από τις εμπλεκόμενες χώρες. Και έρχονται αυτές οι κονσέρβες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με απόλυτη δασμολογική απαλλαγή. Ενώ για τις ε, άλλες προελεύσεις είναι 24% ο δασμός. Αυτό είναι ένα αδιαφυσβήτητο μέτρο το οποίο έχει να κάνει με τις παραδοσιακές παραχωρήσεις που δίνονται στους εταίρους μας από τις χώρες ΑΚΕ για να ευνοηθεί η οικονομική τους ανάπτυξη και δεν υπάρχει καμία δυσκολία και αμφιβολία για τα θέματα αυτά. Οι κανόνες προέλευσης για τον τόνο σαν προτείνουν οι εξή. Αν ο αυτός, οι ηχθείες αυτοί εξάγονται χωρίς μεταποίηση, είτε πρέπει να έχουν αλλιευθεί στα, στα χωρικά ύδατα <clears throat> των χωρών αυτών που εμπλέκονται, όπως είναι η Αγωινέα παραδείγματος χάρη, είτε εκτός των χωρικών υδάτων από ένα πλοίο το οποίο έχει ορισμένη σύνδεση με την χώρα αυτή σημαία, ε, καταγραφή στα νεολόγια και ιδιοκτησία που να αναφέρεται στη χώρα αυτή. Επομένως, για να θεωρείτε μια κονσέρβα, να θεωρείται ότι προέρχεται από μια χώρα, θα πρέπει και είναι λογικό και η πρώτη ύλη της κονσέρβας να προέρχεται από τη χώρα αυτή. Θεωρείται λοιπόν ότι είναι απαραίτητο για αυτό το λόγο το 85% του τόνου που έρχεται στην κονσέρβα να προέρχεται από τη χώρα αυτή το πολύ 15% μπορεί να προέρχεται από άλλες χώρες ώστε να ισχύσει ο κανόνας αυτός ο οποίος οδηγεί σε απολύτη δασμολογική απαλλαγή. Δασμούς 0%. Μετά από το 2008 όμως η συμφωνία αυτή η ενδιάμεση που έτυχε διαπραγμάτευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Παπουασία Νέα Γουινέα επέτρεψε στις χώρες αυτές να παράγουν κονσέρβες οι οποίες θεωρούνται ότι είναι προέλευσης Νέας Γουινέας χρησιμοποιώντας από κάθε λογής προελεύσης πρώτη ύλη με την προϋπόθεση ότι είχαν εκφορτωθεί σε λιμάνια της Νέας Παπουασίας. Αυτή ήταν η μόνη προϋπόθεση. Ο τόνος λοιπόν ο οποίος είχε έτσι εκφορτωθεί θα μπορούσε να έχει αλλιευθεί οπουδήποτε και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Αυτό στρεβλώνει τους κανόνες προέλευσης όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια ριζική και χωρίς προηγούμενο εξαίρεση από τους κανόνες προέλευσης που έχει ολέθρια αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή αγορά ε, κονσέρβας τόνου και στην απασχόληση στον αρμόδιο αυτό τομέα. Από νομική έποψη. Αυτό επιτρέπει <clears throat> μία μορφή ανταγωνισμού που ως εισηγητής γνωμοδότησης και εγώ ίδιος, η εισηγήτρια γνωμοδότηση μάλλον και εγώ ίδιο, διότι θεωρούμε απόλυτα αθέμητη μορφή ανταγωνισμού μετά από την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Στη Νέα Γουινέα έχουν εγκατασταθεί βιομηχανίε μετα... μεταποίηση στη νεα Ουινέα εχουν εγκατασταθει ώστε να μπορούν να εξάγουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε λίγα χρόνια αυτή η χώρα, σε λίγου μήνε ουσιαστικά, έχει γίνει το κέντρο παραγωγή κονσερβών τόνου και ένα παράδεισο κονσερβοποίηση στον Ατλαντικό. Δεν θέλω να σα αναφέρω τι συγκεκριμένε χώρε οι οποίε έχουν αναλάβει τη μεταποίηση. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου μας εξήγησε ότι αυτή η συμφωνία επιτρέπει την βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη της Παπουασίας Νέας Γουινέας. Ως εκ τούτου θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι, να τονίσω ότι καμία από αυτές τις βιομηχανίες δεν ανήκει στην Παπουασία Νέα Γουινέα. Όλες αυτές οι μεταποιητικές βιομηχανίες ελέγχονται από κεφάλαια άλλων ασιατικών χωρών, κυρίως της Κίνας. Και απασχολούν ένα ελάχιστο αριθμό τοπικών εργαζομένων. Γιατί εισάγουν και εργαζόμενους από την Κίνα. Δεν έχουμε ακριβώς στοιχεία για τον αριθμό των εργαζόμενων στις ε, αυτές από την Παπουασία Νέα Γουινέα. Αλλά ακόμα κι αν υπήρχε η δυνατότητα να είναι όλες από την Παπουασία, θα ήταν πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε, αν λάβουμε υπόψη τις αποδοχές των εργαζομένων εκεί, ότι είναι θετικές για την οικονομική ανάπτυξη μια κονσερβοπία, παραδείγματος χάρη από τις Φιλιππίνες και σας δίνω μοναχά ένα παράδειγμα. Απέλησε 400 τοπικούς εργαζομένους πρόσφατα, οι οποίοι διαμαρτυρόντουσαν γιατί δεν είχαν αποδοχές 1 ευρώ την ώρα τουλάχιστον. Καταλαβαίνετε. Έτσι δουλεύουν οι χώρες αυτές. Δεν ε, τίθενται και πολλά ερωτήματα, όποιος δεν συμφωνεί, στον δρόμο. Σήμερα στην Παπουασία Νέα Γουινέα ανθούν οι κονσερβοποίες όπως οι τουλίπες στην Ολλανδία. Βάσει λοιπόν αυτών των συμφωνιών, μια, ένας όμιλος κινέζικων εταιριών έχει καταρτήσει σχέδια που θα οδηγούσαν και σε, στο τέρμα της την παράκτη αλεία στην Παπουασία Νεγουινέα, και θα είχαν πάρα πολύ σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή αυτή. Αυτό θα σημαίνει την ανάπτυξη της μεγαλύτερης ζώνης κονσερβοποίησης τόνου σε όλη την Ασία και τον Ελληνικό, με 30.000 <clears throat> εργαζομένους και 10 βιομηχανίες μεταποίησης του τόνου τη στιγμή που η ανεργία στην Παπουασία Νεγοινέα είναι πολύ ψηλή. Αυτές όμως οι βιομηχανίες θα εισήγαγαν εργαζομένους από άλλες ασιατικές χώρες. Γνωρίζομαι ότι οι κανόνε αυτή προέλευση έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι εμπορικέ παραχωρήσει οι οποίε γίνονται ωφελούν πράγματι του πραγματικού αποδέκτε και δεν θα πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται προ όφελο τρίτων. Αναρωτιόμαστε αν ο στόχο μα είναι η οικονομική ανάπτυξη των Φιλιππινών και τη Κίνα που θέλει να προαγάγει η Κομισιόν με την εξαίρεση αυτή που δίνει στη Νέα Γουινέα. <clears throat> Γιατί ο στόχο είναι η ανάπτυξη τη Νέα Γουινέα, όχι τη Φιλιππίνας το Φιλιππινών ή της Κίνας. Μας λέει εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εισαγωγές κονσέρβας από την Παπουασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αυξήθηκαν ιδιαίτερα μεταξύ του 2006 και του 2009. Αλλά οι, Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίες, ευρωπαϊκές κονσερβοποίες μας λένε κάτι τελείως διαφορετικό. Μας λένε ότι 40.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω αυτής της εξαίρεσης που δόθηκε στην Παπουασία Νεγουίνια. Σε όλη την Ευρώπη 40.000 θέσεις εργασίας. Σε ένα χρόνο θεωρούν ότι η Νέα Γουινέα έτσι θα παράγει πάνω από 200.000 τόνους σε κονσέρβα, ο οποίος θα έρχεται κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι το ίμιση της ισπανικής παραγωγής κονσερβοποιημένων τόνων. Και αυτή η εξαίρεση έχει φυσικά και αρνητικά αποτελέσματα για τα αλλιευτικά αποθέματα. Οι ξένοι στόλοι έχουν ήδη αρχίσει να εποφθαλμιούν τους πόρους τους αλληλευτικούς των χωρών του ειρηνικού. Ενώπιον αυτού του αθέμητου ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή κονσερβοποία, που σας λέω ότι η ευρωπαϊκή κονσερβοποία σέβεται τις προϋποθέσεις για το περιβάλλον, τις κοινωνικές και τις υγειονομικές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ε, αυστηρές, και που επίσης επομίζεται ένα υψηλό κόστος εργασίας, βρίσκεται τώρα η Ευρωπαϊκή Κοσερβοπία σε ένα τεχνητό σύστημα το οποίο βασίζεται σε ε, μη σεβασμό των κανόνων του περιβάλλοντος και των εργασιακών κανόνων. Ενώπιον όλων αυτών, η πρόεδρος μας, κυρία Φράγκα, ζητά εκπεφρασμένα και το σημαίζομαι και εγώ να ανασταλεί αυτή η εξαίρεση το ταχύτερο δυνατό. <clears throat> Μέσα στην πρώτη μεταρρύθμιση της ε, ενδιάμεσης συμφωνίας και φυσικά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τελική συμφωνία η οποία είναι η υποδιαπραγμάτευση. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω αναλάβει το έργο της παρουσίας αυτού του σχεδίου της κυρίας Κάρμεν Φράγα που καταδεικνύει άμεσα τις ανησυχίες που έχουμε εκφράσει όλοι και έχω εκφράσει και εγώ στην έκθεσή μου για την εισαγωγή προϊόντων αλίας και ιχθυοκαλλιέργειας και υποστηρίχθηκε μαζικά από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν μια έκθεση που πραγματικά σοκάρει και έχουμε δύο που θέλουν να σχολιάσουν. Ο κύριος Μαλάνα. Ξεκινάμε τον κύριο Μαλάνα. Κοιτάξτε, όλο αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ ε, σας ερωτώ, έχετε δει ποτέ στις ε, ευρωπαϊκές αγορές ε, μία κονσέρβα τόνου που προέρχεται από την Παπούα, Νέα Γουνέα. Η απάντηση είναι όχι, ούτε από τις Σεϊχέλες. Και εκεί η απάντηση είναι όχι. Όλοι λοιπόν οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι τον τόνο που πουλάνε στην Ευρώπη με τα δικά μας τα εμπορικά σήματα τον ε, κονσερβοποιούν, τον συσκευάζουν σε αυτές τις χώρες. Υπάρχει λοιπόν, ε, υπάρχουν πολλές εισαγωγές από αυτές τις χώρες. Άρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί δεν είναι μόνο οι Κινέζοι που αναπτύσσουν αυτή τη δραστηριότητα, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Εμείς λοιπόν είμαστε εκείνοι που πράττουμε αυτές τις εισαγωγές, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανονισμός που να σχετίζεται με την προέλευση του προϊόντος, κυρίως του συσκευασμένου. Έτσι λοιπόν στην αγορά εμφανίζεται μια πολύ μεγάλη ποσότητα προϊόντων που είναι άμεσα ανταγωνιστικά τα προϊόντα αυτά με εκείνα που παράγουν ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μια Ένα ευρωπαϊκό κλάδο ε, που αλλιεύει στην Ευρώπη και με βάση κριτήρια που συνδέονται με τη δική της την ηθική και δεοντολογία και ε, αυτή είναι ανταγωνιστική με ένα άλλο ε, τύπο ευρωπαϊκής βιομηχανίας που απλά εκμεταλλεύεται τις ε, υπανάπτυκτες χώρες για να παράγει και να συσκευάζει τα προϊόντα της. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό κατ' ουσίαν προκύπτει και από την ε, συμπεριφορά ακόμα και μιας ίδιας εταιρείας, όπου η εταιρεία τα μισά της τα προϊόντα ε, τα παράγει δεοντολογικά σωστά και τα άλλα μέσα από τα κανάλια που σας παρουσίασα. Το θέμα λοιπόν που τίθεται είναι πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση για να δρομολογήσουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση που θα αφορά στην ετικετοθεσία ε, των προϊόντων σε κονσέρβες. Σήμερα στην Ευρώπη είμαστε σε μια κατάσταση όπου μπορεί κανείς να πουλάει ό,τι θέλει σε κονσέρβα χωρίς πάνω στην κονσέρβα να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. Το made in κατόπιν τούτου είναι καθοριστική σημασία. Αυτά λοιπόν που ελέγχθησαν σε σχέση με τους εργαζόμενους, το περιβάλλον, ακόμα και την επιρροή της Κίνας στην Ευρώπη και την Ασία, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η Κίνα επηρεάζει την οικονομία όλων των νοτιοανατολικών χωρών της Ασίας. Το θέμα όμως είναι ότι η δική μας η αγορά δεν θα πρέπει να ανοίξει σε αυτά τα προϊόντα και δεν ανοίγει μέσα από την Κίνα, αλλά μέσα από την Ευρώπη. Άρα δηλαδή θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύστημα όπου θα φύγει το θέμα της προέλευσης των προϊόντων. Ίσως η γνωμοδότηση μπορεί να εμπλουτιστεί ε, και με αυτές τις απόψεις. Εμείς θα το προσπαθήσουμε. Και κατά τα άλλα, επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει το θέμα αυτό ίσως να το συζητήσουμε και με άλλες επιτροπές, γιατί η ετικητοθεσία δεν είναι αποκλειστικό δικό μας προνόμιο. Ε, πάντως ε, όλα ε, τα ψάρια που πολλούνται σε κονσέρβες, σαρδέλες και άλλα θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε εμείς η οποία θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε επί της ουσίας το θέμα αυτό. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μιλάνα, με αυτά που είπε. Δηλαδή υπάρχει πράγματι κανονισμός IEU και εναπόκειται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους ε, δεν προέρχονται από παράνομες ή μη ρυθμιζόμενες πηγές. Ε, το θέμα λοιπόν είναι να εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Και όσον αφορά την Παππούα Νέα Γουινέα, θα πρέπει βεβαίως ε, να εφαρμόζονται οι κανονισμοί του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Επίσης να γίνονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι, διότι αλλιώς θα έχουμε κάθε λόγο Μισό λεπτό λέει ομιλήτρια. μιλήτρια. Δεν, δεν βρίσκω τις λέξεις να τα πω στα αγγλικά, θα πρέπει να περάσω στα σουηδικά. Δυστυχώς δυσκολεύομαι να εκφραστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, στα σουηδικά τώρα. Ε, δεν υπάρχει κανένας ε, λόγος να εγκρίνουμε τις προτιμήσεις αυτές τις δασμολογικές. Και στην Νέα Γουινέα Υπάρχουν ε, Ευρωπαίοι οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτών των ε, εργοστασιακών μονάδων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λόβεν. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Διότι πραγματικά έχω μείνει άφωνος. Σε ό,τι αφορά το 24% που ε, δημιουργήθηκε πανικός και σάλος όταν έγινε μηδέν μέσα σε μια νύχτα αυτός ο εισαγωγικός δασμός. Έχουμε λοιπόν τόνους ψαριών τα οποία πηγαίνουν στην Παπουασία Γουινέα για να κοσορροπηθούν, να σκευαστούν εκεί. Έτσι, δεν εκμεταλλευόμαστε βέβαια μόνο τα τεράστια αποθέματα τόνου, αλλά εκμεταλλευόμαστε και τους εργαζόμενους, τα φτηνά εργατικά χέρια εκεί πέρα. Και επίσης έχουμε και εκατοντάδες απολύσεις, έχουμε πάρα πολύ χαμηλές αμοιβέ και όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο μεταξύ άλλων και τη δική μας μεταποιητική βιομηχανία. Μα ποιος ε, το σκέφτηκε αυτό το πράγμα να το κάνει δηλαδή. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να ακούσουμε μια εξήγηση Γκαρσία Φερέρα από την Κομισιόν πως θα μπορούσε να μας πει κάτι. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω καταρχήν ε, τη συλλογιστική, τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε. ότι είναι καλή ιδέα να δώσω αυτή την ε, παρέκκληση. Είναι μια παρέκκληση στους κανόνες, στους πρότυπους κανόνες προέλευσης. Δηλαδή δεν έχει μειωθεί ο δασμός από το 24% στο 0%. Το 0% αφορά ε, συγκεκριμένα τον ειρηνικό στους κανόνες προέλευσης, στους κανόνες καταγωγής. Πρόκειται για νησιά απομονωμένα, τα οποία βρίσκονται πολύ μακριά, είναι απομακρυσμένα με πολύ λίγες ε, αναπτυξικές δυνατότητες και η έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες ΑΚΕ, τα νησιά του Ειρηνικού έχουν πολύ μικρό αλλιευτικό στόλο που πληρεί τους κανόνες προέλευσης. Δηλαδή, αυτή η δασμολογική προτίμηση που είχαν από το Κοτονού και που μπήκε στο νέο κανονισμό ε, δεν θα τους έδινε κανένα όφελος αν δεν υπήρχε αυτή η παρέκκληση. Εξού λοιπόν και χορηγήσαμε αυτή την παρέκκληση. Και εφαρμόζεται από το 2008 στο πλαίσιο του κανονισμού Market Access Market Access Regulation και το ΕΠΑ μόνο από το 2009 και μετά. Και θέλω να τονίσω ότι, τονίζεται, ότι εφαρμόζεται μόνο για την Παπουασιανεγουινέ γιατί τα ΦΙΤΣΙ δεν πληρούν τα υγειονομικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν μπορούν να εξάγουν. Και δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει ε, την υπογραφή της προσωρινής του συμφωνίας ε, ΕΠΑ, δηλαδή της συμφωνίας, ε, οικονομικής συμφωνίας εταιρικού χαρακτήρα. Τώρα, έχουμε κάποιες πληροφορίες από τη Eurostat εμείς, ε, πληροφορίες που στέλνουν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όλα ε, τα εμπορικά στατιστικά στοιχεία. Βάσει των πληροφοριών αυτών έχει διατηρηθεί το εμπόριο με την Παπουασία Νέα Γουινέα κάτω από το 3% σε ό,τι αφορά τον κορσεβοποιημένο τόνο και σε σχέση με τις συνολικές αγωγές ε, τόνου συσκευασμένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια σημαντική διακύμανση. Πρέπει επίση να έχουμε υπόψη μα το εξή. Οι χώρες αυτές, γιατί μιλήσαμε σήμερα για την παραγωγική τους δυνατότητα, πρέπει να λάβουν υπόψη άλλους παράγοντες που περιορίζουν την παραγωγικότητα. Παραδείγματο χάρη, Έχουμε τον κανονισμό IUU, την αλία IUU. Έχουμε τα υγειονομικά μέτρα, τα ανέφερα. Τι θα πει αυτό. Θα πει ότι πολύ ε, πρώτη οποίοι παράγεται, αλλιεύεται εκεί. Δεν μπορεί να εξαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λιγότερη είναι η πρώτη σε σχέση με αυτό που μπορεί κανείς να φανταστεί. Αυτή, λοιπόν, ε, αυτές οι πρώτες ύλες ε, στην περιοχή αυτή έχει αλληλευτικούς πόρους Παπουασία Νέα Γουινέα, αλλά ουσιαστικά τους ε, εκμεταλλεύονται τα κοσεβοποιία αυτούς τους πόρους άλλων χωρών. Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, θα μπορούσε να γίνει μεταποίηση εκεί, απλά τώρα γίνεται στην Παπουασία Νογουινέα. Θα πρέπει η Παπουασία Νογουινέα να υπερκεράσει πάρα πολλά προβλήματα ανταγωνισμού σε σχέση με τις δύο αυτές χώρες, για να μπορεί να εξάγει τα προϊόντα της στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντικό και αυτό, διότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ ζητούν πολύ υψηλά πρότυπα. Εάν λοιπόν δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα πρότυπα που Νέου, είναι πολύ δύσκολα θα εισχωρήσει σε μια αγορά με τόσο μεγάλη ποιότητα και υψηλή ζήτηση. Και ένα άλλο θέμα το που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα είναι το εξή. Ε, η παραγωγή αυτή από την Παπασία Νέα δεν μπορεί να έρθει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλες αγορέ. Αυστραλία, ΙΠΑ, όπου εκεί υπάρχει επίση μεγάλη ζήτηση συσκευασμένου τόνου. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αντίκτυπο ε, στην Παπουασία Γουινέα, σε ό,τι αφορά την απασχόληση, 5.700 εργαζόμενοι εργάζονται στην Κωσερβοπία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι ντόπιοι, δεν είναι ξένοι, είναι από την Παπασία Νέα Γουινέα αλλά υπάρχει και νομοθεσία που μειώνει στο 7% ε, το ποσοστό των ξένων εργαζομένων στην Παπασία Νέα Γουινέα. Αν εσεί ή ο τομέα, ο κλάδο έχει διαφορετικέ πληροφορίε, σα παρακαλώ να μα τι διαβιβάσετε. Και γιατί σα το λέω αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του παρόντο, ή τέλο πάντων σύντομα, θα εκπονήσει μια έκθεση για ε, την επίπτωση που έχει αυτή η παρέκκληση θα είναι έτοιμη η έκθεση αυτή του χρόνου. Όλε τι πληροφορίε λοιπόν που μπορούμε να έχουμε για να δούμε αν εφαρμόζεται, πώ εφαρμόζεται η παρέκκληση, τι αντίκτυπο έχει και στην Παπασία Νέου Γουινέα και στην Ευρώπη θα είναι πάρα πολύ χρήσιμε πληροφορίε για μα. Και ένα άλλο σημείο το οποίο αναφέρθηκε για τον πιθανό αντίκτυπο στους πόρους ε, στην περιοχή αυτή. Τη διαχείριση την έχει η Επιτροπή του Κεντρικού και Δυτικού Ειρηνικού με πολύ σαφείς αρχές και περιορισμούς. Ήδη λοιπόν πρόκειται για το κατάλληλο πλαίσιο, για να μην έχουμε υπεραλίευση στην περιοχή εκείνη. Είναι μέλος και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την επιτροπή, επομένως μπορούμε και εμείς να ελέγχουμε την εκμετάλλευση των πόρων για να μην υπάρξει υπεραλίευση τους. Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη που πειμένω, αλλά θεωρώ ότι εδώ βασιζόμαστε σε μία λάθος παραδοχή του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα. Αυτό που είπα εγώ ή αυτό που ελέγχει αυτά, το να τα συνδέει κανείς με την εκμετάλλευση ή με την περιθωριοποίηση των πολιτών της ε, παποσία Νέας Γουνέας, το να το πιστεύει κανείς αυτό, αυτό είναι επεσβολητικό για μας, για την ευθεία μας. υπάρχει πράγματι η εκμετάλλευση, αλλά το θέμα είναι ότι τα ψάρια βρίσκονται στα χέρια αυτών των ε, πολιτών και η μεταποίηση στα χέρια των Κινέζων και των Ευρωπαίων. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Και το θέμα αυτό αφορά σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα συσκευασμένα θαλάσσια προϊόντα. Μερικές φορές πρόκειται για τη Νέα Γουνέα, άλλες πάλι ε, φορές πρόκειται για τις Σεχέλες, για οποιοδήποτε νησί που είναι χαμένο κάπου στον Ειρηνικό. Άρα δηλαδή η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει μεγαλύτερη προσοχή τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης και να εισάγει τέτοιου είδους στοιχεία εγγύησης, στοιχεία ίχνη λασιμότητας των προϊόντων για να μπορεί να είναι βέβαιη ότι η αξία του τελικού προϊόντος που διανέμεται στην Ευρώπη έχει πράγματι ε, υπεραξία που προκύπτει από αυτούς τους λαούς. Βεβαίως ε, και την ε, εμπορία αυτών των προϊόντων, αλλά και να ενισχυθούν αυτές οι χώρες. Δηλαδή, ο οικονομικός κύκλος να κλείνει με διαφάνεια και σαφήνεια. Το θέμα που εμείς ε, συζητάμε σήμερα είναι το εξής. Η παραγωγή που φτάνει στην Ευρώπη με απόλυτα ανώνυμη μορφή Πώς μπορεί κανείς να ξέρει ότι πρόκειται για το 3% των προϊόντων. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό. Στην ευρωπαϊκή αγορά δεν αναφέρεται τίποτα που να λέει ονομασία προέλευσης ή την προέλευση. Αυτό το προϊόν από πού προέρχεται και ακόμα και αν είναι μόνο το 3% όμως το 3% της παραγωγής είναι πάρα πολύ υψηλό ποσοστό όταν μιλάμε για ε, ε, ένα προϊόν που διοχετεύεται σε 500 εκατομμύρια κατοίκους. Μιλάμε δηλαδή για ένα προϊόν με μεγάλη οικονομική αξία. Θα πρέπει σε τούτου να γνωρίζουμε τον πραγματικό κύκλο παραγωγής, να κατανοήσουμε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια το ηθικό στοιχείο σε αυτόν τον οικονομικό κύκλο και από την άλλη πλευρά να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής να ενημερώνονται οι καταναλωτές. Γιατί εγώ μιλάω και ως καταναλωτής. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον ο τόνος που αγοράζω ε, στο σούπερ μάρκετ δύο όροφος πιο κάτω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά πόσον ο τόνος αυτός ε, προέρχεται από την Αγουινέ, από τις ΟΧΕΛΕΣ ή από την Ιταλία. Ίσως ε, να διαβάζω πούμε, ότι πρόκειται μια θαυμάσια τελική γαλλική οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, αλλά τελικά ε, αυτό το προϊόν ε, είναι εκείνο για το οποίο συζητάμε σήμερα. Και αυτό δεν μπορεί πια να συνεχιστεί. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό κάνουμε κακό και στους κατοίκους της Νέας Γουινέας και στο ευρωπαϊκό ψάρι και στον ευρωπαίο καταναλωτή. Okay, thank you Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καντέχαν θα ήθελε να παρέμβει και να κλείσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω καταρχήν σε ορισμένα από αυτά τα οποία ελέγχθηκαν. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία εν μέρη με αυτά που είπα προηγουμένως. Οι Ιταλοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό και φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο αυτό το ζήτημα, το συγκεκριμένο είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η προέλευση από τον προϊόντο την ευρωπαϊκά και όχι να εισάγονται από την πίσω πόρτα προϊόντα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την Ευρώπη. Το θέμα των ε, βιομηχανιών μεταποίησης. Τα στοιχεία τα οποία έχω εγώ δεν είναι τα ίδια στοιχεία που έχετε εσείς. Εμένα μου λένε για 10 κινέζικες και φιλιππινέζικες κονσερβοποιίες με 30.000 εργαζομένους. Και όχι 5.700. Νομίζω ότι τα στοιχεία σας είναι ίσως πεπαλαιωμένα γιατί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα οι ασυστιατικές χώρες. Κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα, ένα, μια ευκαιρία, ένα χάσμα το οποίο έπρεπε να εκμεταλλευτούν και κινούνται με εκθετικούς ρυθμούς. Κάθε μέρα αυξάνουν τη δραστηριότητά του. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνείδηση αυτής τη πραγματικότητα και η απάντηση που μας δώσατε εκ μέρους της Κομισιόν δεν θα σας εκπλήξει αν σας πω ότι δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Το ίδιο ισχύει και για τα νησιά πιστεύω. Λέτε για στοιχεία της Eurostat. Εμείς δεν έχουμε πάντως τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε αυτά τα στοιχεία σας για τον αριθμό των κονσερβοποιών στη Νέα Γουινέα, για τον αριθμό των εργαζομένων που είναι αυτόχθονες. Και εμείς οι πληροφορίες που έχουμε πάρει είναι από τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις Παραγωγών Κονσερβοντών και είναι αξιόπιστα στοιχεία. Και σας λέω ειλικρινά, δεν φοβάμαι να το πω αυτό, ότι ουσιαστικά είναι μια δωρεάν παραχώρηση που δίνει σε ορισμένους την ελεύθερη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται προ όφελο ορισμένων και μόνο. Και φυσικά εναπόκειται η απόφαση στην Επιτροπή μας και στη σοφροσύνη των συναδέλφων. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος, κύριε Κάντεκ. Φαίνεται παράξενο ότι ο κύριος ωφελούμενος από όλα αυτά είναι η Κίνα με οικονομική μεγέθυνση 10% όταν η Ευρώπη έχει μεγέθυνση 1%. Η Κίνα και οι Φιλιππίνες επωφελούνται. Πολύ καλό είναι αυτό. Πολύ καλή ιδέα. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι και πάλι στις 12 το μεσημέρι στις 5 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στις 26-27 Οκτωβρίου. Θέλει η Κομισιόν να επανέλθει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ήθελα να διευκρινίσω σε σχέση με τα στοιχεία της Κομισιόν που διαμφισβητήθηκε το αν είναι ενημερωμένο. Οι επιχειρήσεις που έχουν την άδεια να, ε, ε, να εξάγουν από την Παππού Νέα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρεις. Δύο των Φιλιππινών και μία από την Ταϊουάν. 5.700 εργαζόμενους έχουν Υπάρχουν σχέδια τα οποία είναι εν εξελίξη, αλλά χρειάζεται να πάρουν έγκριση για υγειονομικά θέματα, που δεν είναι εύκολο να αποκτήσει κανεί την έγκριση. Η Κομισιόν λοιπόν αυτά τα στοιχεία έχει για τις εισαγωγές που είπατε ότι είναι άλλα στοιχεία. Εμείς έχουμε τα στοιχεία της Eurostat που είναι αυτά που μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη όταν παίρνουν εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα τις καταγράφουν και τις στέλνουν στη βάση δεδομένων της Eurostat. Γι' αυτό είναι πολύ αξιόπιστα αυτά τα αυτά τα στοιχεία για όλα τα προϊόντα και όχι μόνο για την αλληλεία. Άλλα σχόλια θέλετε να κάνετε κύριε Κατέκ? Όχι. Για τα στοιχεία σας λέω ότι διαφυσβητώ προφανώς τα στοιχεία της Κομισιόν και ζητώ από την Κομισιόν με τρόπο άμεσο να αναθεωρήσει αυτά τα στοιχεία, να ξαναδεί ποια είναι η κατάσταση. Σας ξαναλέω αυτό το οποίο σας είπα οι χώρες της Ανατολικής Ασίας κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, εκμεταλλεύονται κάθε εμπορική δυνατότητα με μεγάλη ταχύτητα. Τα στοιχεία σας μπορεί να ίσχυαν πριν από μερικές εβδομάδες ή μήνες, αλλά μην πεπισμένους ότι δεν ισχύουν σήμερα πια και γι' αυτό σας ζητώ να ελέγξετε και πάλι τα στοιχεία σας. Ούτως ή άλλως, η συγήτριά μας, η κυρία Καρμεφράγκα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με αυτή την κατάσταση. Θα δούμε κάποιες ενδιαφέρουσες τροπολογίες λοιπόν. Είναι μια γνωμοδότηση βέβαια. Είναι η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου, η ΙΝΤΑ, η οποία είναι η αρμόδια επί της ουσίας, προθεσμία τροπολογιών 5 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 26 και 27 Οκτωβρίου στην έκθεση ΙΝΤΑ εξωτερικού εμπορίου θα γίνει ψηφοφορία 1η Δεκεμβρίου και θα πάει τον ίδιο το Δεκέμβριο στην Ορομέλεια. Ευχαριστώ λοιπόν και για αυτό το σημείο. Προχωρούμε τώρα στο σημείο 11 συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Λίχτενστάιν. Εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλληλεία. Εισηγητή ήταν ο κύριο Πατικό Γκάλαχερ, ο οποίο δυστυχώ δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Απουσία του κύριου Γκάλαχερ. Θέλω απλώ να σα παραπέμψω στο σχέδιο γνωμοδότησής του που δίνει θετική ε, έχει θετική θέση για την έγκριση της γνωμοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι οι συμφωνίες, οι εν λόγω συμφωνίες δεν σημαίνουν περαιτέρω παραχωρήσεις προς την Ισλανδία και θα πρέπει να είναι σαφές αυτό γιατί ξέρω ότι πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από την διαμάχη που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλανδίας καθώς και των νήσων Φερόε σε σχέση με τα αποθέματα σκόμβρου, θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να εγκρίνουμε τις περαιτέρω αυτές παραχωρήσεις προς την Ισλανδία. Αλλά δεν υπάρχουν πρόσθετες παραχωρήσεις στην Ισλανδία που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν έχει λοιπόν κάποιος από εσά κάποια παρέμβαση, και κάποιο σχόλιο, αν δεν θέλει να λάβει το λόγο η Κομισιόν, σε σχέση με την έκθεση του κ. Γκέλχερ, εγώ προτείνω να καθορίσουμε προθεσμία τροπολογιών για τις 5 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι. Θα ήθελα παρενθετικά να πω ότι υπάρχει και μια τηλεοπτική κάμερα εδώ από το BBC Σκοτίας. Υπάρχει. Και βασικά ενδιαφέρονται για τη συζήτηση περί σκουμβρίου που θα γίνει αργότερα στην Επιτροπή μας. Κυρία Ράιμες, θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Ναι. Μου ζήτησε. Κοιτάξτε, μου ζήτησε ο συνάδελφος να πω κάτι για την ε, γνωμοδότησή του και σχετικά με το ότι η πρόταση αυτή δεν αποτελεί νέα παραχώρηση προς την Ισλανδία όσον αφορά την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Και γι' αυτό λοιπόν ε, συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Αυτό είχα μόνο να πω. Κύριος Χόλνερ από την Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι. Ε, no, thank you, Mr. Chairman. I think uh, there was a rather... Πρόεδρε, ε, έγινε μια μεγάλη συζήτηση και επί της ουσίας δεν έχουμε τίποτα να προτείνουμε. Περιμένουμε να πάρουμε τα σημειώματα από όσους έχουν υπογράψει αυτές τις ε, προσωρινές ε, συμφωνίες και το πρωτόκολλο Ελίας. Προς το παρόν, με δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 5 Οκτωβρίου στις 12 και θα ψηφίσουμε στις 26-27 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΝΤΕ θα είναι στις 9 Νοεμβρίου και μετά ε, το θέμα θα πάει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ε, προχωράμε λοιπόν στην ε, συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Χιλή για τα αποθέματα ξηφίας στο Ανατολικό ελληνικό ε, κοινό. Λείπουν όμως και ο συγητή και η κυρία Φράγκα που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το θέμα αυτό και μας ζήτησαν το θέμα αυτό να αναβληθεί για την επόμενη φορά. Ω εκ τούτου πάμε στο επόμενο θέμα. Α, ε, το επόμενο θέμα είναι η απογευματινή συνεδρίαση. Προχωρήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Ε, είμαι ευγνώμων σε όλους σας γι' αυτό και θα τα ξαναπούμε εδώ για την παρουσίαση της ε, Natura 2000 και για τις ε, συζητήσεις ε, σχετικά με τις τιμές. Θα τα πούμε το απόγευμα στις 3.